κύριος Λαουρέντζιου Ρεμπέκα έχει καταλήψει την ομάδα ε, ΕΝΕΦ από τις 2 Μαρτίου 18 και τώρα είναι με τους μη γραμμένους. Η κυρία Μιράντα έφυγε από την ομάδα Γκούε και προσχώρησε στην ομάδα των Πρασίνων Άλε από τις 2 Μαρτίου 18. Έλαβα από τις ομάδες Ελκ και Πρασίνων